Οι αποδείξεις που έχει συγκεντρώσει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δείχνει ότι τα εγκλήματα μίσους είναι καθημερινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ρατσισμού, ξενοφοβίας, ε, μυσαλλοδοξίας θρησκευτική ή προκαταλήψεις εναντίον της ε, αναπηρίας ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό κάποιου. τα... Μιλάμε για προβλήματα και για βία που στρέφεται εναντίον ολοκλήρων κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υπερασπιστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, και τις μη διακρίσεις. Ε, αυτό είναι δραματικό θέμα. Έχουμε εδώ τον Ιωάννη Δημητρακόπουλο, που είναι προϊστάμενος του Τμήματος Ισότητας και Δικαιωμάτων του Πολίτη. Θα μας παρουσιάσει τα τελευταία συμπεράσματα του οργανισμού του για το θέμα αυτό. Κύριε Δημητρακόπουλε, αν μπορείτε να μας παρουσιάσετε το θέμα, θα ήταν καλό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρουσιαστώ εδώ και να συζητήσουμε τα εγκλήματα μίσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η διεύθυνσή μου παρουσίασε την τελευταία έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2013, προειδοποίησε ότι τα στοιχεία ε, που συγκεντρώσαμε δείχνουν τα εγκλήματα λόγω ρατσισμού, ξενοφοβίας, και διάφορων μυσαλλοδοξιών, ε, εξτρεμιστικής ιδεολογίας στην πολιτική και δημόσια συζήτηση, ε, εθνικές διακρίσεις ε, στην εκπαίδευση, στη στέγαση, σε διάφορους τομείς, υπάρχουν παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βασίζεται σε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο οργανισμός μας σε διάφορα διάφορα χρόνια για διάφορες μορφές εγκλημάτων μίσους εναντίον μεταναστών, μειονοτήτων, θρησκευτικών, πολιτικών, εθνικών κτλ. Εμείς κάναμε τις έρευνες αυτές. Επίσης έχουμε αναλύσει επίσημα στοιχεία. Πρέπει να τονίσω ότι μόνο τέσσερα κράτη-μέλη ε, συλλέγουν πλήρη στοιχεία για Φιλανδία, Ολλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο για τα εγκλήματα μίσους. Άλλες Άλλα 12 ε, δημοσιεύουν κάποια δεδομένα, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουν τους μηχανισμούς καταχώρησης και αποτύπωση των εγκλημάτων μίσους. Λόγω των αναποτελεσματικών επίσημων στοιχείων και για να δώσουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αξιόπιστα και συγκρίσιμα ε, στοιχεία, ούτω ώστε να προωθήσουμε πολιτικέ που να βασίζονται σε στοιχεία και να δώσουμε νομικέ απαντήσει, ο οργανισμό μα έκανε πανευρωπαϊκέ έρευνε. Ε, 23.500 ε, χιλιάδες ε, άτομα ε, ερωτήσαμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, επιλέξαμε τυχαία 22.000 ε, Ρωμά για να μας δώσουν πληροφορίες για 84.000 84 νοικοκυριά σε 11 κράτη-μέλη. Επίσης, η επισκόπησή μας πάνω σε ομοφιλόφιλους άνδρες και γυναίκες, φιλομεταβατικούς και ενδοφιλικούς, ε, αφορούσε όλα τα κρατημέλη. Τρεις χιλιάδες ήταν τα άτομα που επιλέξαμε να, πάρουμε, να ρωτήσουμε. Μιλούσαμε, τους ρωτούσαμε για τις εμπειρίες τους. Τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, που είναι και τα πιθανότερο να πέσουν θύματα αυτών των εγκλημάτων, έχουν δυνατότητα να μιλήσουν ε, κατά την ανάλυση μας, ε, αυτά δίνουν και αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές, ούτως ώστε όσοι προωθούν τις πολιτικές να καταλάβουν καλύτερα την κατάσταση και να λάβουν στοχευμένη και αποτελεσματική δράση. Κυρίες και κύριοι, οποιοδήποτε μπορεί να είναι θύμα ε, εγκλήματος μίσου. Στην πραγματικότητα αυτό το φαινόμενο κυρίως επηρεάζει τις πιο ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία μας. Δεν πρόκειται να σας ε, πνίξω στα νούμερα, αλλά θα σας δώσω κάποια παραδείγματα από τις έρευνές μας που δίνουν τις επιπτώσεις, δείχνουν τις επιπτώσεις των εγκλημάτων αυτών. Όπως σας είπα, αυτή η πανευρωπαϊκή έρευνα που έγινε για τους μετανάστες και, και τους Ρώμα ε, δείχνει ότι ο ένας στους πέντε ε, Ρωμά και Αφρικανούς από την Υποσαχάριο Αφρική δείχνουν ότι το ένα λοιπόν στους πέντε ε, έχουν πέσει θύμα τέτοιου εγκλήματος τα τελευταία τον τελευταίο χρόνο. Ένας από τους δέκα μουσουλμάνους επίση που απάντησαν ε, θεωρεί ότι είναι θύμα τέτοια παρενόχληση στους τελευταίου 12 μήνες. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση ε, έρευνας, ούτως ώστε να προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία για να αξιολογήσουμε την επίπτωση των ε, ευρωπαϊκών και εθνικών νομικών και πολιτικών απαντήσεων τα τελευταία χρόνια. Η έρευνά μας για τις έρευνες που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο δείχνει ότι κατά μέσο όρο ε, ένα στους πέντε Εβραίους ε, έχει πέσει θύμα φυσικής βίας ή παρενόχληση σοβαρής, μόνο και μόνο γιατί είναι Εβραίος. Επίσης οι ομοφιλόφιλοι κατά 26% έχουν πέσει θύματα ε, κάποια στιγμή μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια και το νούμερο φτάνει το 35% για τους φιλομεταβατικούς. Αυτά τα νούμερα δείχνουν απλώς σε ποιο βαθμό τα εγκλήματα αυτά πλήττουν αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Αυτό είναι, αυτό είναι ισχυτικό και πρέπει να το διορθώσουμε. Μην ξεχνάμε ότι τα εγκλήματα μίσου επηρεάζουν όχι μόνο τα θύματα, αλλά τις οικογένειές τους και τους φίλους τους. Ε, προκαλεί φόβο και αβεβαιότητα. Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της ε, έρευνάς μας για αυτά τα εγκλήματα δείχνουν ότι όσο διαφορετικοί και αν οι άνθρωποι ως προς την εθνική τους προέλευση, τι τους του, το στυλ ζωή του και στην εθνικότητά τους επηρεάζονται από το, φόρο, από το φόβο τέτοιων ε, αδικημάτων. Φόβο ότι θεωρούνται πως ανήκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα, φόβο ότι μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο και φόβο ότι τα μέλη της οικογένειάς τους και αυτά μπορούν να πέσουν θύματα. Στην πρόσφατη έρευνα που κάναμε για τους Εβραίου, περίπου το 50% είπαν ότι ανησυχούν για τον εαυτό τους, τις οικογένειε τους ή τους φίλους τους, ότι μπορεί να πέσουν κάποια στιγμή θύμα ενό ενός τέτοιου εγκλήματος. Ε, και λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για να μην γίνουν θύμα ενός τέτοιου εγκλήματος. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι αναγκαίο όμω σε μια ελεύθερη δημοκρατική ε, κοινωνία όπου συμμετέχουν όλοι. Όσοι είπαν ότι ανησυχούν πω μπορεί να πέσουν τέτοια θύματα, ε, είπαν κατά 76% ότι αποφεύγουν να φορούν, να, μεταφέρουν κάτι που να τους ε, ταυτοποιεί με την ε, ευρεότητά τους. Ε, επίσης, το 1 τέταρτο περίπου από τους ε, ανθρώπους που απάντησαν είπαν ότι δεν πηγαίνουν σε εκδηλώσεις εβραϊκές γιατί δεν αισθάνονται ασφάλεια. Από την έρευνά μας για τους ομοφιλόφιλους, ίδια αποτελέσματα. Το 50% είπαν ότι δεν κρατιούνται χέρι-χέρι με τον σύντροφό τους, ίδιου φίλου, γιατί φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα παρενόχλησης. 50% επίσης των ατόμων είπαν ότι αποφεύγουν συγκεκριμένους τόπους, γιατί φοβούνται ότι μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων, μόνο και μόνο γιατί είναι ομοφιλόφιλοι άντρες ή γυναίκες, φιλομεταβατικοί κτλ. Αυτά τα εγκλήματα παραβιάζουν σαφώ τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη ζωή και στην ακεραιότητα ενός ατόμου. Ο φόβος αυτού του εγκλήματος παραβιάζει το θεμελιώδης ε, δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια, δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε ελεύθερα και ανοιχτά και αυτό είναι απαράδεκτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου περιγράφεται στις συνθήκες ως ε, κοινωνία όπου πλουραλισμός, η έλλειψη διακρίσεων, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη κτλ. Ενταξύ ανδρών και γυναικών υπάρχουν. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια εγκλήματα. Η τα εγκλήματα αυτά δείχνουν ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικά ε, νομικά μέτρα και πολιτικέ. Ε, ο οργανισμό μα ε, καλωσορίζει το σχέδιο έκθεση τη Επιτροπής σα για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καταδικάζει το ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, την ομοφιλοφοβία, την ξενοφοβία, τη βία κατά των μεταναστών, θρησκευτικών μειονοτήτων, εθνικών ομάδων κτλ. Ε, οι λόγοι είναι διαφορετικοί κάθε φορά. Ε, συχνά όλα αυτά δείχνουν ότι τα άτομα επίσης, ε, πρέπει να προσθέσω μάλλον τα άτομα ε, με αναπηρίες μπορούν να είναι θύματα και θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων υποφέρουν. Είτε γίνονται θύματα λόγω της εθνικής τους προέλευσης, της θρησκείας τους, του χρωματός τους, του φίλου τους, του σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της αναπηρίας τους. Έχουμε λοιπόν ε, αναφέρει κάποια παραδείγματα στη γνωμοδότησή μας για την απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και είπαμε ότι όταν προστατεύουν τα δικαιώματα των θυμάτων, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους λόγου των προκαταλήψεων και όλα τα χαρακτηριστικά ε, που προβλέπει το άρθρο 21 της ε, Χάρτας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και να καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Από τις έρευνές μας ε, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ε, ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις μειονοτικές ομάδες δεν γνωρίζουν αυτή την νομοθεσία. Ε, δεν ξέρουν ότι μπορεί να προστατευτούν. Αυτοί που ανήκουν σε μειονότητες λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν νόμοι και ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Ε, αυτό θα βοηθούσε ούτω ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην δικαιοσύνη και να αναφέρονται, να καταγγέλλονται αυτά τα εγκλήματα στην αστυνομία. Για την καταχώρηση αυτών των αδικημάτων, αυτών των ε, αδικημάτων ε, η έρευνά μας δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό ε, στην αναφορά και καταγγελία αυτών των εγκλημάτων. Τα περισσότερα άτομα που ανήκουν σε τέτοιες μειονότητες δεν προσφέρουν στην αστυνομία. Κυρίως γιατί, όπως λένε, δεν πιστεύουν ότι κάτι θα κάνει η αστυνομία ή θα αλλάξει κάτι με το να τα καταγγείλουν. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των διοκτικών αρχών για να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά του είναι προφανώ ανησυχητική. Καλωσορίζουμε λοιπόν τα συμπέρασματα του Συμβουλίου τη 5η και 6η Δεκεμβρίου του 2013 για το έγκλημα μίσου, που καλεί την υπηρεσία μα να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στι προσπάθειέ του να ενθαρρύνουν την καταγγελία και να γίνεται σωστή καταχώρηση των εγκλημάτων αυτών με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής των καλών πρακτικών. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά την διάσκεψη που κάναμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα τον Νοέμβριο του 2013 ε, θα συνδιοργανώσουμε τέλος Απριλίου ένα σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ίδια θέματα, τόσο ώστε να προωθήσουμε αυτό το σημείο. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές και διαπιστώνουμε με ανησυχία ε, κάποιες δημοσκοπήσεις ε, και σφιγμομετρήσεις στα κράτη-μέλη που δείχνουν ότι αυξάνεται το εκλογικό σώμα των εξαμιστικών πολιτικών ε, κομμάτων που ανοιχτά μιλάνε κατά των μειονοτήτων. Τον περασμένο μήνα δημοσιεύτηκε μία έκθεση από εμά για δύο κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Ουγγαρία, ε, ως ε, περιπτώσεις όπου αξίζει να συζητήσουμε τις προκλήσεις λόγω ρατσισμού, ε, μυσαλλοδοξίας και εξτρεμισμού. Εστίασε αυτή η έρευνα στις δύο χώρες, αλλά κατέληξε σε μία σειρά συμπερασμάτων, πολύ ευρεά συμπεράσματα, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εγκλήματα. Ε, καταρχάς, μπορούμε να αναπτύξουμε εθνικές στρατηγικές κατά του ρατσισμού ε, και της ε, μυσαλλοδοξίας ε, με συνεργασία διαφόρων εταίρων, με την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, να αυξήσουμε την, το επίπεδο κατάρτισης της αστυνομίας και τη δυνατότητα της, των εισαγγελικών αρχών να αντιμετωπίσουν περίπλοκα εγκλήματα μίσους. Τελειώνοντας, μια άλλη σημαντική διάσταση στα εγκλήματα αυτά είναι κάτι που συχνά ξεχνάμε. Το έγκλημα αυτό όχι μόνο μια ουσιαστική πρόκληση ε, στις ε, βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωση, που είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη και η ε, ισότητα, αλλά ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη και μια κοινωνία που να λαμβάνει υπόψη όλου και που είναι η καρδιά της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ε, αν υπάρχει μυσαλλοδοξία και τέτοια εγκλήματα, ε, τα μέλη δεν μπορούν να ζήσουν, τα μέλη της κοινωνίας αυτής δεν μπορούν να ζήσουν και να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους. Ο χαμένος δεν είναι μόνο το άτομο, αλλά ολόκληρη κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Δημητρακόπουλε για την ε, εξαιρετικά λεπτομερή και ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας. Θα δώσω τώρα το λόγο του συναδέλφους, αρχίζοντας από την κυρία Κόντς πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Τα στοιχεία που μας παρουσιάζετε μας προκαλούν ανησυχία. ανησυχία. Θα μπορούσατε να μας πείτε πόσα άτομα έχουν την εντύπωση ότι είναι θύματα διακρίσεων. Κάνοντας σύγκριση των ε, στοιχείων που έχετε, μπορείτε να μας πείτε πόσα στοιχεία έχετε και εκθέσει ανάλογα με τη χώρα, διότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ε, ε, διαφορές, κυρίως μεταξύ των ατόπων που φοβούνται ότι κάποια στιγμή θα πέσουν θύματα μιας ε, διακριτικής μεταχείρισης. Και πάλι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας σε κάποιες ε, συζητήσεις που είχαμε. Αφενός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν ζητούσε τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δει ποιε είναι οι απειλές που υφίστανται τα, η αμφιφιλική, η διαφιλική, η κτλ για να δούμε τι ακριβώς γίνεται στις χώρες αυτές. Και περιμένουμε στοιχεία τα τελευταίους μήνες. Δεύτερον, η νοδηγία για τις ε, οριζόντιες διακρίσεις. Ε, ξέρουμε ότι ήδη έχει αρχίσει η όλη διαδικασία στο Συμβούλιο, δεν έχει υπάρξει όμως μεγάλη πρόοδος, ότι κάποιες χώρες ανθίστανται. Νομίζω ότι μπορείτε να βοηθήστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΑ για να προχωρήσουν κάποια στοιχεία εκ μέρους Επιτροπής, ώστε να αυξηθεί η πίεση και να μπορέσει να δημοσιεύσει αυτό τον οδικό χάρτη η Κομισιό και να προωθηθούν μετά οι συζητήσεις στην ε, Συμβούλιο για την οδηγία αυτή κατά των διακρίσεων. Επίσης αναφέρεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι πολιτικές επιπτώσεις καθώς και το πολιτικό ε, ε, κλίμα. Αναφέρατε δύο ε, περιπτώσεις που μελετήσατε με εξτρεμιστικά δεξιά κόμματα, τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, το ένα αντίστοιχο κόμμα στην Ουγγαρία και τώρα από ό,τι ε, λένε, λέει ο αγγλικός τύπος, ο εκπρόσωπος αυτού του κόμματος στην Ουγγαρία θέλει να επισκεφτεί την Αγγλία. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα και κίνδυνος. Εάν κάποιος πάει σε μια άλλη χώρα από τη δική του Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει εκστρατεία αντιευρωπαϊκή και μιλήσει κατά των ευρωπαϊκών αξιών. Είναι λοιπόν πολιτικό καθήκον όλων μας κατά κάποιο τρόπο να υψώσουμε τη φωνή μας και να είμαστε απόλυτα σαφή σε αυτή την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογέ και να πρέπει πραγματικά να εξηγήσουμε σε όλους ποια είναι τα πραγματικά και θεμελιώδη ε, δικαιώματα, οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ανθυρή η κατάστασή μας γενικότερα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε ε, ενδιαφέρον ε, το οποίο είναι απαραίτητο για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία Κόντσα, κυρία Σίπελ. Ja, vielen Dank. Ähm, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάτι που αναρωτιέμαι κάθε φορά όταν κοιτάμε τα νούμερα. Από την έκθεση αυτή γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Έχουμε ήδη πρόβλημα διότι τα κριτήρια για την καταγραφή τέτοιων ε, πράξεων είναι διαφορετικά και αν κάποια κράτη-μέλη δεν υποβάλλουν κανένα στοιχείο τότε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι υψηλότερα από αυτά που συγκεντρώνονται Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία, από... γιατί από κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχουν στοιχεία. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν παίζει ρόλο στη... στους συλλογισμούς σας το εξής. Από την έναρξη της κρίσης έχουμε δει αύξηση του ε, δεξιού εξτρεμισμού πράξεις βίας και ακούμε συνεχώς σε δημόσιες συζητήσεις ότι αυτό οφείλεται στην κρίση και μόλις ξαναυπάρξει ανάπτυξη θα ε, τελειώσουν όλα αυτά. Εμένα αυτό μου φαίνεται απλοϊκό. Ακούγεται σαν φυσικό φαινόμενο, θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Φυσικό φαινόμενο είναι, αύριο θα λάμπει πάλι ο ήλιος και έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Για μένα αυτό είναι υπερβολικά απλοϊκό. Τίθεται το θέμα για μένα Υπάρχουν έρευνες, μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών. Μπορούμε να δούμε πόσο τολμηροί, πόσο δραστήριοι είναι οι πολιτικοί και ε, άνθρωποι από άλλους φορείς και τι επιτυχία έχουν ε, τέτοιες δραστηριότητες, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πέντε χρόνια μέχρι να ξαναυπάρξει ανάπτυξη θα πρέπει σε δύσκολους ε, καιρούς να προασπιστούμε τις αξίες μας. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να αναφέρω, διότι είπατε ότι δεν γίνεται μήνυση σε περίπτωση κάθε τέτοιας ε, πράξης μίσους. Είναι, υπάρχει το γενικό αίσθημα ότι ούτως ή άλλως δεν βοηθάει, δεν έχει νόημα ή οφείλεται αυτό στο ότι οι αρχές δίωξης προσπαθούν να βρουν τους δράστες αλλά δεν έχουν αρκετούς πόρους, αρκετό δυναμικό για να διασφαλίσουν την προστασία αυτού που υποβάλλει τη μήνυση. Υπάρχουν θετικά παραδείγματα σχετικά με το πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά ώστε να υποβάλλεται μήνυση σε περίπτωση κάθε εγκλήματος μίσους. Merci, Madame Sipel. Et maintenant, la parole est à... Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάσης ήταν το λόγο. Ε, ja, dank u, ε, mevrouw de, voorzitter. Ε, Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οποιαδήποτε πράξη μίσους πρέπει να είναι πράξη αξιόπινη με αυστηρή ποινή για οποιαδήποτε, για οποιοδήποτε ε, είδους αδίκημα ή έγκλημα. Μας παρουσίασε κάποια στοιχεία ο κύριος Δημητρακόπουλος, σύμφωνα με το οποίο είδαμε ότι πάρα πολύ συχνά οι κυβερνήσεις αριστεράς και ομάδες της αριστεράς χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα για να περιχαρακώσουν το δικαίωμα έκφρασης. Ακούσαμε να αναφέρουν διάφορα επιχειρήματα και οι σοσιαλιστές και οι δεξιοί. Η κυρία Γκένς ανέφερε δύο πολιτικά κόμματα, τα οποία όμως μας με ενοχλούν εμένα διότι ακούμε μόνο να γίνεται λόγος για κόμματα τα οποία είναι κατά του, του, χαρ, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πολύ συχνά μας προσάπτουν ότι είμαστε κατά των ευρωπαϊκών αξιών. Αυτά διότι επικρίνουν κάποιοι την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο λειτουργία της και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιούνται κατά κάποιο τρόπο κάποιες μελέτες σαν και αυτές που μας παρουσιάζονται σήμερα και εγώ θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου και το λέγω ευθέως τον κύριο Δημητρακόπουλο αυτό δεδομένου ότι υπάρχουν άτομα τα οποία διαπράττουν εγκλήματα μίσους και τους δίνουμε κάποια στοιχεία. Στην σελίδα 13 του που αναφέρεται στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να μας δώσετε εμάς περισσότερες πληροφορίες για τις μειονοτικές ομάδες οι οποίες διαπράττουν τέτοιου είδους εγκλήματα μίσους. Διότι αν δούμε ποιες είναι οι αντισημιτικές πράξεις ή ρατσιστικές αν θέλετε κατά των ε, ομοφιλοφίλων βλέπουμε ότι στην Ευρώπη κυρίως τέτοιου είδους ε, πράξεις βίας διαπράττονται από μουσουλμάνους στην Ευρώπη. Άρα είμαστε λίγο ασαφείς σε σχέση με αυτό το θέμα το οποίο είναι μια αλήθεια που δεν μας ε, βολεύει κατά κάποιο τρόπο να παρουσιάσουμε. Και πολλές φορές κάποιοι παρουσιάζονται ως θύματα ενώ θα ήθελα εμείς να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή πώς μπορούν να διαπράξουν εγκλήματα μέσως και κάποια άτομα τα οποία είναι από μειονοτικές ομάδες. Ο κύριος Μπρονξ πρώτα απ' όλα. Ε, τα εγκλήματα μίσους είναι ένας ε, όρος ε, που διατυπώθηκε πρώτη φορά στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν είναι η καλύτερη εξαγωγή. Γενικά θεωρείται βίαιο έγκλημα το οποίο έχει ω κίνητρο την κατηγορία από την οποία προέρχεται το θύμα. Ε, αυτό θεωρείται ε, επιβαρυντικός παράγοντας ε, στο στο δικαστήριο. Ε, τώρα το αν είναι χειρότερο το έγκλημα επειδή μου κλέβουν το πορτοφόλι επειδή είμαι ένας ηλικιωμένο λευκός και από ότι εάν είναι από, ε, ε, από, από, άλλα κίνητρα αυτό μπορεί να συζητηθεί. Όπως και να έχει πολλά εγκλήματα μίσους που έχουν να κάνουν με θρησκεία ή πολιτική ε, διαπράττονται από μέλη μειονότητας εις βάρος μέλων, ε, μελών πλειονότητας. Ε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον Κρίς ε, Ντόναλντ, έναν ε, νέο λευκό, ο οποίος ε, σκοτώθηκε από μια συμμορία ασιατών στη Γλασκόβη. Ή τον Λί Ρίγμπι που πρόσφατα αποκεφαλίστηκε στο Λονδίνο από δύο μέλη φιλετικής μειονότητας που ήταν και μουσουλμάνοι. Αυτά λοιπόν είναι θύματα ε, εγκλημάτων μίσους. Ε, υπάρχουν και πολλοί διευθύντες καταστημάτων των οποίων ε, τα καταστήματα καταστράφηκαν στο Λονδίνο. Επίσης του Στίβεν Λόρις η δολοφονία ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο τότε διότι ήταν εξαίρεση. Ε, αλλά οι επιθέσεις κατά ανθρώπων λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού ήταν ε, πολύ σπάνια πριν ε, τρεις ή τέσσερις δεκαετίες. Η εξαίρεση όμως είναι οι μουσουλμανικές περιοχές του Λονδίνου. Γίνονται επιθέσεις κατά ανθρώπων λόγω ιδεολογίας. Νομίζω ότι και αυτά είναι κλίματα μίσους. Είχαμε μία συνέντευξη τύπου μετά τις ε, ευρωεκλογές του 2009 και επιτέθηκαν ε, εναντίον μας ε, με μεταλλικά βεράκια από μια ομάδα της οποίας ο σπόνσορας ήταν ακόμα και ο David Cameron. Και η αστυνομία δεν προσπάθησε καν να παρέμβει. Ακούσαμε σήμερα το πρωί από την πλατφόρμα ε, ομιλία μίσους. Ακούσαμε και το κοινό να αναφέρει όρους ε, ακροδεξιός, ε, ρατσιστής ε, κλπ. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα ύπουλο μήνυμα προς τον κόσμο να, ακούσει, να, σταματήσει να ακούει και απλά να μισεί τον ομιλητή. Ε, υπάρχει πολύ μικρό βήμα ανάμεσα στις λέξεις αυτές και τις πράξεις μίσους τις οποίες αναφέρθηκαν νωρίτερα όλες οι πράξεις βίας θα πρέπει να καταδικάζονται άσχετα από το ποιος είναι ο δράστης, άσχετα από το ποιο είναι το θύμα και ποιο είναι το κίνητρο. Θα πρέπει όλοι να το λέμε αυτό. Sorry, uh, just, just one sentence to Mr. Clay, who... Μία πρόταση προς ε, τον ε, κύριο που ανέφερε το όνομά μου. Πρόκειται για παρανόηση. Δεν μιλούσα εγώ για τον ευρωσκεπτικισμό γενικά, μιλούσα για κόμματα τα οποία αμφισβητούν τις ε, θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω και να σχολιάσω τις δηλώσεις σα. Ε, καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν συνταγματικέ διαφορές και διαφορές ε, ως προς ε, τους ορισμούς στα διάφορα κράτη-μέλη που δυσκολεύουν την συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων πάνω στα εγκλήματα μίσους. Ωστόσο, αναμένουμε το κάθε κράτος μέλος εντός του δικού του συνταγματικού πλαισίου, ε, εντός του δικού του εθνικού νομικού ε, πλαισίου να συλλέγει επαρκή δεδομένα. Κατά την εξέταση των παραδειγμάτων που ανέφερα, εάν κοιτάξουμε και άλλες χώρες, διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός ε, συμβάντων που Εξετάζουμε μάλλον τον αριθμό συμβάντων ε, που αναφέρονται στην αστυνομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις αυτές είναι εγκλήματα μίσους. Ε, μπορεί να έχει κανείς δεκάδες χιλιάδες ε, συμβάντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι εγκλήματα μίσους. Οι αρχές δίωξης, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να δούνε ποια από αυτά είναι κλίματα μίσους και ποια όχι. Αλλά για τους πολιτικούς και σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουν προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουν οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. Η συλλογή λοιπόν στοιχείων πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς εργαζόμαστε με αυτό το στόχο, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που ζητούν από μας να προωθήσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου, την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. Θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, θα διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και θα δούμε εάν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα καλύτερο σύστημα αναφοράς των εγκλημάτων μίσους. Αναφέρθηκε το θέμα της κρίσης και το βαθμό που ε, αυτή οδηγεί σε εξτρεμισμό θα διαπιστώσετε και το λέμε αυτό στην έκθεσή μας ότι δεν υπάρχουν παρόμοιες εξελίξεις σε ε, άλλες χώρες που πλήττονται από την κρίση όπως είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ωστόσο, για τις δύο χώρες που αναφέραμε σημειώνουμε ότι επί πολλά χρόνια, ήδη από τη δεκαετία του 90, το Συμβούλιο της Ευρώπης και Κάποιοι άλλοι διεθνείς ε, φορείς χτύπησαν συναγερμό σχετικά με την κατάσταση των μειονοτήτων και, την, και τον ρατσισμό. Δεν είναι λοιπόν κάτι που εμφανίστηκε το 2008-2009. Εάν εξετάσει κανείς ε, την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης ε, του κράτους ε, θα πρέπει να κάνει κανείς την διάκριση στην ε, αντίδραση αντιμετώπιση σε επίπεδο πολιτικών δηλώσεων, να λέει κάποιος δηλαδή ότι υπάρχει μηδενικό περιθώριο ανοχής σε διάφορες μορφές ρατσισμού, αλλά αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από δουλειά σε επιχειρησιακό και τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να συνοδεύεται από δουλειά σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Όσον αφορά τους λόγους που δεν αναφέρονται τα εγκλήματα αυτά, ε, οι περισσότεροι άνθρωποι στις ε, μελέτες που σας ανέφερα, είτε πρόκειτο για ε, Εβραίους, άλλες μειονότητες ή άτομα ΛΟΑΔ, από προηγου... οι περισσότεροι θεώρησαν ε, ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή. Έτσι λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και ε, χάνει το κουράγιο του. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα μείγμα βέλτιστων πρακτικών. Ε, θα ήθελα να αναφέρω μία που εδώ και δύο χρόνια εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για προσπάθεια οικοδόμηση εμπιστοσύνη ανάμεσα στι κοινότητε, ε, τι ε, αρχέ επιβαλή του νόμου ε, και τη δημιουργία νέων τρόπων να αναφέρονται τα εγκλήματα μίσου. Λέγεται Facing Facts το πρόγραμμα αυτό και έχει καταφέρει να συνεργαστεί με εβραϊκέ κοινότητε και κοινότητε ΛΟΑΔ, λεσβιών ομοφυλοφίλων, αμφιλοφίλων και διεμφυλικών και γίνεται τώρα προσπάθεια να συνομιλήσουν και με μουσουλμανικέ κοινότητε όπως σας είπα, εγώ πιστεύω ότι το έγκλημα μίσους αφορά όλους μας. Ε, είναι ένα σύννεφο που ε, γράμεται πάνω από την κοινωνία μας και αφορά όλους μας. Επίσης, ε, δεν εξετάζουμε εμείς περιπτώσεις δηλώσεων μίσους, ασχολούμαστε μόνο με τα εγκλήματα μίσους. τα εγκλήματα μίσου, ο σωστός όρο είναι εγκλήματα που οφείλονται σε προκαταλήψεις. Δηλαδή έχουν να κάνουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Ε, οι εγκληματίε μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε κοινότητα, μπορεί να είναι οποιοδήποτε εγκληματία που ζει σε κάποια χώρα. Υπάρχει όμω ε, διαφορά ανάμεσα στο γενικό έγκλημα και το έγκλημα που οφείλεται σε προκαταλήψει. Και εξετάσαμε τις περιπτώσεις ε, Αυτόν που διαπράττουν τα εγκλήματα. Δεν θυμάμαι τα ακριβή νούμερα, αλλά ε, στις έρευνές μας υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτούς που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά και θα διαπιστώσετε ότι ε, τα πρόσωπα αυτά ήταν και ε, άτομα από την ίδια κοινότητα μειονοτήτων, άτομα από άλλες κοινότητες μειονοτήτων ή άτομα από τον γενικό πληθυσμό που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για ένα συγκεκριμένο ε, έγκλημα μίσους. Επίσης ε, στην έρευνά μας ε, στις εβραϊκές κοινότητες είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί ισορροπές στα διάφορα στη Γαλλία και το Βέλγιο. Κυρίως περιγράφονται μουσουλμάνοι ως εξτρεμιτές και θεωρείται ότι είναι εγκληματίες στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε τους εξτρεμιστές ή χριστιανούς εξτρεμιστές. Είναι ωστόσο σημαντικό να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των εγκλημάτων μίσους, όπως είπα και πριν, δεν επηρεάζονται μόνο οι συγκεκριμένες μειονότητες. Είναι τα θύματα, αλλά από την άλλη το σύνολο της κοινωνίας επηρεάζεται, διότι ε, μειώνεται η κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ, κύριε Δημητρακόπουλε. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο τώρα, εάν συμφωνείτε. Περνάμε στο σημείο 20. Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της Ατιμία και των δημοκρατιών της Κώστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα και Παναμά από την άλλη, ως αφορά το, το άρθρο 49, παράγραφος 3. Η κυρία Ρενάτε Βέμπερ είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει γίνει μια πρώτη παρουσίαση της κατάστασης και της πρόθεσης που επιδιώκουμε με αυτή την έκθεση. Επομένως δεν χρειάζεται να ξανακάνω από την αρχή την παρουσίαση. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι εταίροι μας και οι φίλοι από τις χώρες Κεντρικής Αμερικής περιμένανε αυτή τη συμφωνία να τεθεί σε ισχύ Δέκα χρόνια. Και έχουμε τη δυνατότητα τώρα να το κάνουμε. Η ΛΥΜΠΕ είναι υπεύθυνη μόνο για το άρθρο αυτό που αφορά την αμοιβαία επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών. Όμως χρειάζεται αυτό να εσωματωθεί στη Συμφωνία για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία. Επομένως, η πρότασή μου με την έκθεση είναι να δώσουμε την συγκατάθεσή μας, τη σύμφωνη γνώμη μας, στη συμφωνία αυτή και ελπίζω ότι δεν θα υποβληθεί καμία τροπολογία. Θα δούμε όμως. Πιστεύω επίσης, επίσης ότι θα ψηφίσουμε σύντομα στη ΛΥΜΠΕ και στην Ολομέλεια. Ελπίζω μάλιστα πριν το τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Μια και είναι πραγματικά σημαντικό να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Je Μόλις έφτασε η Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Κύριε Σούλτιν, θέλετε να πείτε κάτι. Δεν είναι ακόμη κανένας παρόν εκ μέρους της Επιτροπής. Ναι, ναι, κάποιος έχει φτάσει. Έφτασε, μάλιστα. Uh, yes, thank you. Good afternoon. Um, ES, e uh, Πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό το να τέθει σε εφαρμογή αυτή η συνθήκη της ε, χώρες της Κεντρικής Αμερικής έγιναν οι σχετικές ε, ε, επικυρώσεις για θέματα επαναξιολόγησης επανήλθε η όλη έκθεση στην Επιτροπή προς έγκριση αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όταν πρόσφατα επισκέφθηκε τις χώρες και τις Αμερικής ο κύριος Μπαρόζο. Είπαν όλοι οι αρχηγοί κρατών πόσο σημαντικό είναι αυτό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τις θέσεις μας. Τώρα βασιζόμαστε στην συνθήκη του 1993. Η συμφωνία σύνδεσης θα αντικαταστήσει ε, την παρούσα όταν θα ε, τελειοποιηθεί, όταν ε, θα εγκριθεί. Ελπίζουμε λοιπόν ότι όλη η διαδικασία θα προχωρήσει αρκετά σύντομα. Θέλει κανένας άλλος συνάδελφος να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Τυχεροί είστε κυρία Βέμπερ. Θα ήθελα να μου πει η γραμματεία πότε θα γίνει ψηφοφορία, διότι ε, δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Πότε θα ψηφίσει η Επιτροπή μας, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 30 Ιανουαρίου στις 12, ε, έγκριση 12 και στην δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί η έκφραση στο Στρασβούργο. Σχεδόν σίγουρες οι ημερομηνίες αυτές που δίδω. Άρα ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας και για τώρα σας ευχαριστώ όλους.